ευκαιρίες καθώς και τους τίτλους αυτών των νομικών πράξεων. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο σχέδιο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο εγκρίθηκε από την διάσκεψη των Προέδρων στις 16 Μαΐου, έχει διανεμηθεί σε όλους και δεν υπάρχει καμία αλλαγή για την σημερινή ημερήσια διάταξη, για τη Τρίτη και την Δετάρτη. Οι προφορικές ερωτήσεις για την Κολομβία και το Περού θα μεταφερθούν από την Πέμπτη στην Τρίτη το απόγευμα. Επίσης η οικονομική βοήθεια για τις τρίτες χώρες θα περάσει από την Τετάρτη στην Πέμπτη. Για την Τετάρτη δεν υπάρχει καμία προτινόμενη αλλαγή. Αν δεν υπάρχει και από δική σας πλευράς καμία συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης ημέρησης διάταξης, μπορούμε να αποχωρήσουμε. Κύριε Λούλινγκ, κύριε Πρόεδρε, εκπλήσωμε γιατί βλέπω ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτού του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ημερήσια διάταξη αυτής της εβδομάδας. Είχαμε κάνει μια πρόταση για μια προφορική ερώτηση για την κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό απερίφθη. Και για άλλη μια φορά θα μιλήσουμε για το θέμα της ομοφοβίας. Πραγματικά υπάρχει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνει το θέμα αυτό στην συνθήκη. Γιατί λοιπόν διαρκώς αγνοούμε προτεραιότητες που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την ε, γεωργία και διαρκώς ε, εστιάζουμε την προσοχή μας στην ομοφοβία. Κυρία Λούλινγκ, ξέρετε ότι οι επικεφαλής των ε, πολιτικών ομάδων είναι αυτοί που αποφασίζουν και το θέμα της ε, ομοφοβίας ε, βεβαίως έχει προταθεί και βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Ελπίζω να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα άλλα θέματα που έχουν προταθεί στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Όντι. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται σε επίπεδο ανεπισήμου συμβουλίου και κανονικά ακόμα και όταν είναι ανεπίσημα τα συμβουλία ο Προεδρεύων θα πρέπει να έρθει εδώ και να αναφερθεί στα συζητήσεις αυτές. Διαρωτώ λοιπόν αν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει προσκληθεί και τι εξηγεί το ότι δεν ήρθε εδώ να αναφερθεί στο τι έγινε στο Συμβούλιο το οποίο επαναλαμβάνω ήταν ανεπίσημο βέβαια. Τι να σας πω, εδώ με δυσκολεύεται κύριε Όντι. Έχετε δίκιο, τον καλέσαμε, δεν ξέρω γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση, αλλά έχετε δίκιο. Ξέρω ότι ο κύριος Βαν Ρον Πόι διστάζει να έρθει, αρνήθηκε να έρθει, απαντώντας ότι δεν έχει κάποιες ανακοινώσεις να κάνει. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο ότι ο κύριος Βαν Ρόνποϊ καλό θα ήταν να μας ενημερώσει, να συνεννοηθεί μαζί σας για το τι θα πρέπει να ανακοινωθεί στην διάσκεψη αρχών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και έχω την εντύπωση ότι για τόσο σημαντικές ε, συναντήσεις ε, στο Συμβούλιο βεβαίως και θα έπρεπε προηγουμένως ο κύριος Βαν Ρομπόι να έρχεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Εντάξει. Θα ενημερώσω για την ε, άποψη του Κοινοβουλίου και βεβαίως θα προσπαθήσω να είμαστε παρόντες και στην τελική φωτογραφία. Λοιπόν, όσον αφορά την ημερήσια διάταξη δεν υπάρχουν αλλαγές, γι' αυτό και θα περάσουμε στο πρώτο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης, έκθεση Μπουζουτήλ. Πρόκειται για τον πίνακα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα Είναι μεγάλη κουβέντα για την ανάπτυξη και το πώ θα δώσουμε κάποια όθηση στι οικονομίε τη Ευρώπη, ώστε